Επίσης θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι σε συνεργασία και μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου υπέγραψα μια νομοθετική πράξη της συνήθους νομοθετική διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 78 και πρόκειται αυτό να δημοσιευθεί στα πρακτικά. Και τώρα έχουμε